Oui. Oui, Ok. Bonsoir, chers collègues. Si vous permettez, on va commencer. Παρακαλώ συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε τη συνεργασία μας. Μπορώ να σας πω ως μέλος του Ευρωκοινοβουλίου εδώ και μια δεκαετία ότι η αίθουσά μας ως Επιτροπή των Γυναικών δεν είχε ποτέ τέτοια πληρότητα. Κυρίζω την έναρξη της συνεδρίασης και καλωσορίζω όλα τα μέλη για αυτήν την ε, πρώτη μας ε, συνάντηση. Yeah. Καταρχήν θα εκλέξουμε τον την Πρόεδρο και μετά έναν έναν τους αντιπρόεδρους. Θα ήθελα να παρατηρήσω ότι κατά διάρκεια της συνεδριάσεως δεν έχουμε διαθέσιμη διερμηνία προς τα Μαλτέζικα. Η κυρία Φων Στόρκ, παρακαλώ, έχετε ζητήσει το λόγο. Ε, ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ μία ερώτηση αναφορικά με την διαδικασία που θα ακολουθεί. Θα ήθελα να γνωρίζω εάν οι ομάδες προτίθενται να εργαστούν με βάση ένα σύστημα DONT. Δηλαδή θα τηρήσουν το σύστημα DONT ή όχι. Μπορούμε να ζητήσουμε χωριστές ψηφοφορίες ε, για την α ή β θέση. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να εφαρμόσουμε το σύστημα DONT. Νομίζω ότι οι προσωπικές απόψεις δεν πρέπει να υπερισχύσουν εδώ. Δεν ε, χρειάζεται να έχουμε ιδεολογικές ε, θέσεις ε, και να λάβουμε τις αποφάσεις με τρόπο καθαρά δημοκρατικά, δηλαδή μέσω του συστήματος DONT. Θα ήθελα να γνωρίζω τι πιστεύουν οι υπόλοιποι συντονιστές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Φωνστόκ. Δεν νομίζω ότι τώρα μπορεί να διεξαχθεί συζήτηση. Χρειάζεται να συνεχίσουμε τη συνεδρίασή μας, αλλά όπως είπατε οι υποψήφοι θα είναι πάντα υποψήφοι οι οποίοι επιλέγονται με τα βάση το σύστημα του. Εγώ μπορώ να ελπίζω το σύστημα αυτό θα τηρηθεί και στην συνεδρίαση αυτή. στόχος της συνεργασίας μου είναι η συγκρότηση του Προεδρείου με την εκλογή της, του, της Προέδρου και με την εκλογή τριών-τεσσάρων αντιπροέδρων. Σύμφωνα με τον κανονισμό μετά από τις εκλογές θα εγκρίνουμε το ε, χρονοδιάγραμμα των συνεργάσεων της Επιτροπής Γυναικών για το 2014 αλλά και το γλωσσικό προφίλ και μετά θα περάσουμε στις ε, αναγγελίες της Πρόεδρου. Επειδή δεν είναι παρόν όλα τα τακτικά μέλη στη σημερινή συνεδρίαση θα σας ε, αναφέρω τα ονόματα των αναπληρωματικών μελών που μπορούν να ανικαραστήσουν τους ε, τακτικούς. Η κυρία Βαν Χέλτ, η κυρία Κωνσταντζα Κρύπ, ο κύριος Άντερ η κυρία Σαμπίν Βερχάιεν, η κυρία Μόνικα Χολμάιερ, η κυρία Λάρα Κόμι, κυρία Μπριάννα Βορτσάν, κυρία Μαρίτα Ουσκόκ, ο κύριος Μαρκ Ταραβέλα, κυρία Μπιλμπάου Μπαραντίκα, κυρία Ιντβέλτ και ο κύριος Στεφάν Εκ. Θα ήθελα να σας πω πως σε... αν υπάρχει κάποια αλλαγή σε ό,τι προανέφερα στα ονόματα, τότε τα κράτη οι πολιτικές ομάδες θα πρέπει να το αναφέρουν πριν από την έναξη των ψηφοφοριών. Η γραμματεία έχει ετοιμάσει όλους τους καταλόγους ε, των παρόντων. Για να είναι έγκυρη η ψηφοφορία θα πρέπει να επαληθεύσουμε την απαρτία. Απαιτείται το 1 των μελών, άρα χρειάζεται τουλάχιστον 9 μέλη να είναι παρόντα στην συνεδρίαση. Προτού να προχωρήσουμε στην εκλογή του Προέδρου, νομίζω πως ε, θα πρέπει να ελέγξουμε το ηλεκτρονικό σύστημα. Ε, φυσικά χρειάζεται να υπάρχουν δύο υποψήφοι τουλάχιστον, διότι αν υπάρχει μία υποψήφιος ε, θα την εκλέξουμε διαβοής. Ε, οι παρακάτω υποψηφιότητες έχουν γίνει δεκτές για την Προεδρία. Μία μόνο είναι η υποψήφια Πρόεδρος, κυρία Ιράτσε Γκαρτσία Πέρες από τη Σοσιαλιστική Ομάδα. Υπάρχουν άλλες υποψηφιότητες για την Προεδρία της ε, Επιτροπής Γυναικών. Όχι, άρα ψηφίζουμε διαβοή. Συμφωνείτε. Συγχαρητήρια κυρία Γκαρσία Πέρες. Συνεργαζόμαστε εδώ και μια δεκαετία με την κυρία Γκαρσία Πέρες, άρα με ιδιαίτερη χαρά την υποδέχομαι στην Προεδρία. Eh, Αγαπητοί Αγαπητέ συνάδελφοι, να σας ε, ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη που δείξατε στο πρόσωπό μου. Ελπίζω πως η εργασία και η συνεργασία με όλους τους συναδέλφους ε, της Επιτροπής θα οδηγήσει στην βελτίωση των σχέσεων ανδρογυναικών και των δικαιωμάτων. Ελπίζω λοιπόν να προχωρήσουμε με την συνεργασία σας. Σας ζητώ υπομονή ευθύς εξ αρχής. Χρειάζεται κάποιος χρόνος για να συνηθίσουμε στον τρόπο εργασίας ε, της Επιτροπής μας. Και τώρα θα περάσουμε στην εκλογή των αντιπροέδρων. θα αναφέρουμε τα ονόματα των ε, αναπληρωματικών ε, για το ΕΛΚ Γκαλπέλτ, Grip, Ντέλη, Βερχάγεν, Αν Holmeyer. Αν Λαρακόμε. Λυπάμαι για την προφορά. Θα βάλω το δυνατά μου λοιπόν για να βελτιωθώ για την ομάδα Άλτε, Νταντσίλα. Κοχ, Αν Μαρταραβέλα. Por ε, el grupo ALDE, Για την ομάδα ALDE, Μπιλμπάλ Βαρντίκα. Αν Σοφία Ιμπέλ. Por el grupo de e. Για την ομάδα GUE, Στέφαν Εκ. Αν δεν έχουν γίνει αλλαγές, να περάσουμε στην εκλογή της πρώτη αντιπροέδρου διαπιστώνοντας ε, πως υπάρχει ε, απαρτία. Περάσουμε λοιπόν στην εκλογή της πρώτης αντιπροέδρου. Υποψήφισα από πλευρά ΕΛΚ έχουμε την κυρία Ματέρα. Εάν δεν υπάρχει άλλος ή άλλη υποψηφιότητα για την πρώτη αντιπροεδρία. Διαβόης λοιπόν να εγκρίνουμε την υποψηφία της Ματέρα. Sí, por favor, la señora Stork. Παρακαλώ, κυρία Στόρκ. Ευχαριστώ πολύ είχα το εξής ε, ερώτημα. Κατά πόσο είναι δυνατό οι συντονιστές αν θέλουμε να διατηρήσουμε τους τέσσερις ε, ε, αντιπροέδρους ή αν θέλουμε να αλλάξουμε το σύστημα αυτό και να έχουμε λιγότερους αντιπροέδρους. Θα ήθελα να έχω μια απάντηση λοιπόν σε σχέση με την άποψη των συντονιστών για αυτό το θέμα. bueno, no podemos entrar ahora a un debate al Δεν νομίζω ότι μπορούμε να συζητήσουμε τώρα για το θέμα αυτό. Πιστεύω πρέπει να συνεχίσουμε την ψηφοφορία για τις αντιπροεδρίες όπως έχει προβλεφθεί. Αν υπάρχει τώρα κάποια παρατήρηση που θέλετε να κάνετε, μπορείτε να την κάνετε. Περνάμε λοιπόν στην εκλογή της δεύτερης αντιπροεδρίας. Από την ΚΟΕ προτείνεται η κυρία Ινές Ζούμπερ. Είναι εδώ παρούσα. Υπάρχει κάποιο άλλο υποψήφιο, κάποια άλλη υποψήφιος. βοή λοιπόν η κυρία Ίνες Ζουμπέρ εκλέγεται δεύτερη αντιπρόεδρος. Παρακαλώ. pasamos a la elección de la tercera vice... Τρίτη αντιπροεδρία από τους σοσιαλιστές. Προτείνει κυρία Μπλινκεβιτσιούτε. Συγγνώμη για την προφορά μου. Si no hay ninguna candidata más, eh, por Αν δεν υπάρχει άλλος υποψήφιος, εγκρίνουμε την κυρία Μπλινκεβιτσιούτε δια ω τρίτη αντιπρόεδρο. Ελάτε να καθίσετε παρακαλώ. Και τώρα έχουμε την εκλογή της τέταρτης αντιπροεδρίας από την ε, ομάδα ECR έχουμε την υποψηφιότητα της κυρίας Φων Εστόρκ. Κύριε Ταραμπέλα, θέλετε να πείτε κάτι προηγουμένως. Να απαντήσω στο ερώτημα που έθεσε η κυρία Βον Στόρκ. Πράγματι μπορεί να υπάρξει αίτηση μυστικής ψηφοφορίας για, την, για κάποια αντιπροεδρία. Το σύστημα DONT είναι σεβαστό μεν, αλλά μπορεί πάντα κανείς να ζητήσει μια ψηφοφορία χω, ε, χωριστή. Εγώ ζητώ μυστική ψηφοφορία για την κυρία Μπέατρις Φανστόρ που είναι τέταρτη αντιπρόεδρος. Υποψήφια για τέταρτη αντιπρόεδρος. La colega Win, Win Servisca. Perdón. Να εκφραστώ κατά της απόφασης. Με εκπλήσει πως μετά από τις τέσσερις ψηφοφορίες που είχαμε κανένας δεν έφερε αντίρρηση και σε αυτή την ξαφνική, ξαφνικά σε αυτή την περίπτωση κάποιος ε, προβάλλει μορφή. Νομίζω ότι εδώ πέρα πρόκειται για διάκριση σε βάρος της δικιάς μας υποψηφίου και αυτό αντιβαίνει στου κανόνες της διπλωματίας ε, και της δημοκρατίας. Sí, eh, la colega... Καλώς. Πίρτερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Εγώ υποστηρίζω το αίτημα για μυστική ψηφοφορία, λέει η κυρία Μπέρντερ. Εδώ στο Κοινοβούλιο πάντα οι ευρωβουλευτές έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν όπως επιθυμούν. Και εδώ η υποψηφιότητα αυτή είναι τέτοια που θα τα καλύτερα να ψηφίσουμε. Θα ήταν πιο εύκολο να ψηφίσουμε πρώτα απ' όλα αν θα έχουμε μυστική ψηφοφορία ή όχι. Αυτό διανατάσσεως της χειρό θα έλεγα. Πρόεδρος, ο κανονισμός προβλέπει ότι μπορεί να ζητήσει κάποιος τη διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας, η οποία λαμβάνει στη συνέχεια χώρα, εφόσον τη στηρίξουν το έτοιμο αυτό, δηλαδή έξι ευρωβουλευτές. Από ό,τι βλέπω υπάρχει αυτή η στήριξη, άρα δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε περισσότερο, να περάσουμε να δούμε κατά πόσο θα κάνουμε τη μυστική ψηφοφορία. Παρακαλώ λοιπόν τους συναδέρφους με τις ηλεκτρονικές τους κάρτες να ψηφίσουν. Η κυρία Σινάνσκα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θέλω να εκφράσω εδώ την έκπληξή μου που η Επιτροπή αυτή, η οποία αναφέρεται στην ισότητα, η οποία έχει να κάνει με την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, που θέλει και την ισότητα ευκαιριών, τώρα κάνει διάκριση σε βάρος ενός μέλους της. Δεν θα ακολουθήσουμε δηλαδή την ίδια διαδικασία όπως είχαμε ακολουθήσει και στις προηγούμενες ψηφοφορίες. Δεν έχει νόημα αυτό. Ναι, θέλουμε να είμαστε ελεύθεροι, βεβαίως, και θέλουμε να ψηφίζουμε ελεύθερα, ανοιχτά. Και ψηφίστε κατά άμα δεν θέλετε. Τι πρόβλημα έχετε. Πρόεδρος, δεν θέλω να ανοίξουμε και πάλι τη συζήτηση. Επαναλαμβάνω ότι στον κανονισμό προβλέπεται η δυνατότητα να ζητήσει κανείς μυστική ψηφοφορία για έναν υποψήφιο στην Αντιπροεδρία. Αφού το προβλέπει ο κανονισμός λοιπόν θα αποφασίσουμε θα το κάνουμε ή όχι. Θα έχουμε μυστική ψηφοφορία ή όχι. Χρειάζονται έξι τουλάχιστον που θα στηρίξουν το αίτημα για μυστική ψηφοφορία. Οπότε ψηφίζουμε επί του αιτήματο αυτού για μυστική ψηφοφορία. Α, γίνεται και διανατάσσεω της χερός. Λοιπόν, ποιο συμφωνεί για μυστική ψηφοφορία τώρα. Να σηκώσει το χέρι. Ευχαριστώ. Πάνω από έξι βλέπω. Συνεπώ, η ψηφοφορία θα γίνει μυστικά για την θέση του τετάρτου αντιπρόεδρου της Επιτροπής μας. Eh, Οπότε, έχετε τις κάρτες σας. Στο μηχάνημα παρακαλώ, βάλτε το στο μηχάνημα. Τέσσερα σημαίνει υπέρ της κυρίας. Άσπρο σημαίνει αποχή και κόκκινο σημαίνει κατά. Ναι, κυρία Σαμπόσκα, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ξέχασα τη δικιά μου κάρτα σε κάποια άλλη επιτροπή. Μπορείτε να υπολογιστε και τη δικιά μου την ψήφο. Εγώ θα ψηφίσω ανοιχτά. Όχι μυστικά. De acuerdo. Abrimos la... Καλώς. Αρχίζουμε την ψηφοφορία. Μπορείτε να ψηφίσετε τώρα. Esperamos la 30. Esperamos. Esperamos a Campúa. 31. Podemos cerrar. Eh, Cerramos el voto. Πέρα τη ψηφοφορία. 13 ψήφοι υπέρ, 17 κατά και μία αποχή. Συνεπώς η κυρία Φον Στόρκ δεν εξελέγει στη θέση της τετάρτης αντιπροεδρίας της Επιτροπής μας. El Συνεπώς, η τέταρτη αυτή αντιπροεδρία θα περιμένει μέχρι την επόμενη συνεδρίασή μας για να έχουμε ξανά υποψηφιότητες κλπ. Καλώ. Καλώς. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης που είναι η έγκριση των ημερομηνιών που θα συνεδριάσουμε μέσα στο υπόλοιπο 2014. Είναι ο κατάλογος με τις ημερομηνίες αυτές, απλώς πρέπει να εγκρίνεται το χρονοδιάγραμμα δηλαδή. Συμφωνούμε? Καλώς, εγκρίνεται λοιπόν. Και το επόμενο σημείο έχει να κάνει με το γλωσσικό προφίλ. Θέλει κανείς κάτι να πει εδώ, υπάρχει κάποιο θέμα. Bueno, entonces lo damos para probado. En cuanto a... Εγκρίνεται και αυτό. Και έρχομαι στις ανακοινώσεις τώρα ε, της Πρόεδρου. Πρόκειται για το σχέδιο προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2015 και το χρονοδιάγραμμα το σχετικό. Η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι 24η Ιουλίου. Μέχρι τότε μπορείτε να υποβάλλετε τροπολογίες. Και η έγκριση θα λάβει χώρα στην Επιτροπή στις 13 Σεπτεμβρίου στην Επιτροπή μας μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Λοιπόν, 24 Ιουλίου είναι η προθεσμία για να υποβάλλετε τις τροπολογίες σας στον προϋπολογισμό και 3, 3, Σεπτεμβρίου, συγνώμη, 3 Σεπτεμβρίου θα εγκρίνει η Επιτροπή μας το σχέδιο προϋπολογισμού. Ευχαριστώ και θα τα πούμε στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας.